επιτροπή του οι τέσσερις αιτήσει και ε, άρσης ασυλίας του κυρίου Χέρν να θεωρηθούν απαράδεκτες. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στις 11 και 12 Φεβρουαρίου επικέρωσε την εντολή των κυρίων Μπέργκερ, Τσιριτάφη, Μέριου, Μανόλε, Ματούλα, Ναζάριση, Τόνεν, Αντόκι και Ντάντζιλα αφού έλεγξε τις εντολές αυτές βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισμού μας και ομόφωνα προτείνει να θεωρηθούν έγκυρες οι εντολές αυτές. Υπάρχουν αντιρρήσεις, εάν όχι έχουν επικυρωθεί οι εντολές των ηρημένων συναδέλφων. Η Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων αντιμετώπισε το θέμα της εφαρμογής του άρθρου 47 του